Καθίστε παρακαλώ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Το τελευταίο θέμα της ημερής διάταξης είναι ενημέρωση σχετικά με την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε από τις, ε, στην ε, Κωνσταντινούπολη πρόσφατα. Καλωσορίζω την ε, κυρία Εύα Καηλή που είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας μας. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την δυνατότητα να ενημερώσω τις 11 και τους συναδέλφους DNAT για την 22η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΣΤΟ που έγινε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Φωτίγκα και τον κύριο τον Στρεύσκη, τον κύριο Βανόρντεν και τον κύριο Νικολάη που, ήταν, που συμμετείχαν στην αποστολή. Η συνέλευση ε, πραγματοποιήθηκε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τέσσερις μήνες μόλις μετά την, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος και λίγες μέρες πριν από την υπερψήφιση ενός σημαντικού ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο που, που όπως γνωρίζετε καταδίκασε τα δυσανάλογα κατασταλτικά μέτρα που έχει λάβει η Τουρκία ως απάντηση στο πραξικόπημο και που οδήγησε στο προσωρινό πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Υπήρξαν λοιπόν πολύ έντονες συζητήσεις για το, την απόπειρα πραξικοπήματος, ιδίως με, τους, ε, ε, με την κυβέρνηση και το στρατό της Τουρκίας που ε, επέκριναν πολύ στεναρά το, το γεγονός ότι οι σύμμαχοι επέδειξαν απροθυμία αρχικά να καταδικάσουν την, το πραξικόπημα και για το γεγονός ότι έχει ε, φορτωθεί υπερβολικές ευθύνες η Τουρκία για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών από τη Συρία. Να τονίσω ότι ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να γίνει ολόκληρη ένα τεράστιο hot spot προσφύγων αν η Τουρκία αποφασίσει να τους επιτρέψει να εισέλθουν στην Ένωση, ενώ πολλοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι τα πάντα συμβαίνουν με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές στην ε, χώρα. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίθηκαν σοβαρά από τους ε, ε, Τούρκους ε, όσον αφορά τα, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, όσον αφορά την καταπολέμηση της, τρομοκρατίας και την απόπειρα πραξικοπήματος. Επίσης, ε, ε, ασκήθηκε κριτική από την, πλευρή, από την πλευρά μας στην Τουρκία για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τους πραξικοπηματίες. Οι, οι, οι τουρκικές αρχές ε, τονίστηκε στη, ε, ε, ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο μια στρατιωτική συμμαχία, αλλά μια συμμαχία η οποία υπερασπίζεται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και πολλοί από εμά τόνισαν και την ανάγκη διαφύλαξης της ελευθερίας λόγου και έκφρασης στη χώρα. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα όπως το Ισλαμικό κράτος, η Ουκρανία, η Ρωσία, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, γιατί πολλοί άνθρωποι πλέον συνδέουν την ε, προσφυγική κρίση με τον ΝΑΤΟ και το καλούν να αναλάβει δράση. Και άλλα ζητήματα συζητήθηκαν, η μετάβαση στο Αφγανιστάν, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η καταπολέμηση της διαφοράς. Ε, ο Γενικός Γραμματέας Στόλτεμπεργκ υπογράμμισε τις ε, δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, μας έδωσε δηλαδή κάποιες ε, πληροφορίες, ιδίω όσον αφορά την ανάπτυξη τεσσάρων ταγμάτων στις χώρες της Βαλτικής και απέστειλε ένα μήνυμα ενότητας του ΝΑΤΟ και μια καλύτερη κατανομή των βαρών, ιδίω του, του προϋπολογισμού, όπως η Πολωνία και η Ελλάδα που πληρώνουν 2%, αλλά ε, άλλες χώρες ε, ε, δεν έχουν επιτύχει ή δεν θέλουν να επιτύχουν τον συγκεκριμένο στόχο. Επίσης, χαιρέτησε την όρμη που υπάρχει το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και ε, υπενθύμησε και την κοινή ε, διακήρυξη που υπεγράφει μεταξύ των διοργανώσεων των τον ε, Ιούλιο στη Βαρσοβία αλλά και τα συμπεράσματα που, του Συμβουλίου που είχαν εγκριθεί δύο μέρες νωρίτερα. Εμείς θέσαμε ερωτήσεις στον Γενικό Γραμματέα. Εκείνος χαιρέτησε την συνεργασία μεταξύ των διοργανώσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και ε, τόνισε ότι οι κοινή ε, ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας δεν θέλουν να αποτελέσει ένα αντινάτο, θέλουν να είναι μια διαδικασία συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική προς τη συμμαχία. Παρ' όλα αυτά τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι ικανότητες, οι επιχειρησιακές της συμμαχίας και της αύξησης των δαπανών. Όσον αφορά το έγγραφο που σας ε, διένυμα, σας ε, ε, έχω συμπεριλάβει και κάποια στοιχεία για την πολύ έντονη συζήτηση, κάτι που ήταν ασυνήθιστο ε, για κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, όμως συνέβη στην Κωνσταντινούπολη. όλα αυτά θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους τα μέλη της ΔΙΝΑΤ. Νομίζω ότι έχουμε πλέον ενισχύσει σοβαρά την ορατότητά μας σε αυτή την κοινοβουλευτική συνέλευση. Να ευχαριστήσω επίσης τη Γραμματεία για την παρουσία της και για την υποστήριξη που μας παρήχε την παρακολούθηση όλων των ε, εργαστηρίων. Τέλος, ε, εκλέξαμε και νέο πρόεδρο. Ο, νέο, ο κύριος Πάολο Άλλη ε, από την Ιταλία εξελέγει για μονοετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Είναι και καλός μας φίλος και μου φίλος και θα συνεργαστώ μαζί του το συντομότερο δυνατόν, ίσως και από τον Ιανουάριο και έπειτα, ε, στο πλαίσιο των συναντήσεων DINAT. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστούμε κυρία Καλή, λέει η Πρόεδρος, για την ανασκόπηση αυτών των ε, γεγονότων. Ήρθε στη σωστή ώρα. Ήταν πολύ χρήσιμο. να γίνει αυτή η συνάντηση της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Ήταν σημαντική η σύμβολη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις εκεί συζητήσεις. Και εγώ να ευχαριστήσω βεβαίως τη Γραμματεία και τους άλλους συνεργάτες μας. Όλοι που βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Μας βοήθησαν πραγματικά. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Κύριε Γκόμες, μήπως θέλετε κάτι να προσθέσετε. Uh, Θα ήθελα να ρωτήσω τι συνέπειες είχαν οι δηλώσεις Τραμπ όσον αφορά την πίστη των μελών της συμμαχίας. Κύριε Γιώργη, θέλετε και εσείς το λόγο. Ναι. Κύριε Καλή, θέλετε να απαντήσετε. Uh, ναι, ναι. Βεβαίω και Αναφέρθηκε αυτό και πολλοί συνάδελφοι ανησυχούν για το μέλλον της συμμαχίας. Και άλλοι, όπως οι γενικός βέβαια, πιστεύουν ότι πρόκειται να έχει μέλλον η συμμαχία. Και συμφώνησαν σε εκείνο το σημείο που ο Τραμπ είπε ότι όλοι θα πρέπει να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας και να συμβάλλουμε στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Να μην θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει όλου να μας βοηθάει χωρίς όλοι να συμμετέχουμε στα οικονομικά. Γιατί έχουμε τέσσερι χώρε μόνο που συμμετέχουν στον συμφωνηθέντα προπολογισμό. Και αν θέλουμε να διευρυνθούν οι επιχειρήσεις στα σύνορα ή στην ε, Μεσόγειο να μας βοηθήσει στο προσφυγικό, να βοηθήσει στη Συρία. Ε, για να γίνουν αυτά θα πρέπει και να βοηθούμε οικονομικά. Πάντως, πήγαμε στην οσυντών λίγες μέρες μετά, πήγαμε την αντιπροσωπεία για τη σχέση με τη ΣΥΠΑ, μιλήσαμε με γερουσιαστές και μέλη του Κογκρέσου, ακόμα και οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν έχουν σε κάθε εικόνα για το τι μέλη γενέστε. Δεν μπορούν να σχολιάσουν, δεν ξέρουν από ποιον θα επηρεάζεται ο πρόεδρος. Ε, θεωρούν ότι θα υπάρχει επιρροή από τον αντιπρόεδρο και δεν ανησυχούν για την ύπαρξη του ΝΑΤΟ ή για τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Είναι πάντως ε, ανήσυχοι και για τη συμφωνία με το Ιράν επίσης ε, θα υπάρξει κάποια ένσταση και αυτό θα ζητηθεί την επόμενη φορά. θα υπάρξει δυσκολία με τη νέα κυβέρνηση. Και άρα θα πρέπει η Ευρώπη να έχει αποκτήσει μια δική της στρατηγική. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο της ημέρας της Ευχαριστούμε την αντιπροσωπεία μας. Πότε αυτή την σημαντική για το Κοινοβούλιο Αποστολή. Κυρίε και κύριοι, στις 25 Ιανουαρίου είναι η επόμενη συνεδρίασή μα 25 και 26 Ιανουαρίου. Οπότε σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Να ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Καλύτερες ευχές μας. Και σε εκείνους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους και σας ευχαριστώ. Γιατί όλη αυτή την ε, χρονιά δουλέψαμε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Εκτιμούμε πάρα πολύ τη βοήθειά σας. Ε, Βεβαίω και η γραμματεία μας βοήθησε πάρα πολύ. Κύριε Σόντερ, και εσείς τις καλύτερες ευχές μας.